Καλό σας απόγευμα. Αρχίζουμε με μια μικρή καθυστέρηση δεδομένου τη συνεχής τη συζήτηση του Προέδρου και να δούμε τι γίνεται στη ημέρα διάταξη. Η ε, παράκληση του κυρίου Σούστα βάσει του κανονισμού 115 το θέμα των εμπορικών διαπραγματεύσεων με το Μερκοσούρ θα προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη. Από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννικ, θέλεις να μιλήσεις όσον αφορά την ε, ανακοίνωση. Έχουμε βρει λύση, άμα θέλεις μπορείς να μιλήσεις λίγο επ' αυτού. Όπως αναφέρατε μόλις, Πρόεδρε, θέλουμε να μιλήσουμε για την έκθεση της, uh, early Και γι' αυτό θέλουμε να μπει στην ατζέντα. Γιάννικ, Κοίταξε, θα το βάλουμε, θα το προσθέσουμε μεταξύ του θέματος 5 και 6. Βεβαίως υπάρχει το ρίσκο να μην είναι παρούσα η Κομισιόν, αυτό το δέχεσαι. Ωραία, δεν έχετε άλλες αντιρρήσεις, υποθέτουμε. Θεωρούμε την ημερήσια διάταξη εγκεκριμένη και προχωρούμε στο θέμα 2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 26ης 27 Νοεμβρίου. Θεωρούμε ότι τα πρακτικά εγκρίνονται εκτός αν υπάρχουν σχόλια στο τέλος της συνεδρίασης. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο εκτός από τα τμήματα που είναι και κλεισμένων των θυρών έχει διανεμηθεί η μερίσια διάταξη. Αν ενδιαφέρεστε για κάτι συγκεκριμένο, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία όσον αφορά τώρα την ε, συμμετοχή στι συνεδριάσεις TLD. Ο κύριος Μορέιρα βέβαια, μιλώ εκ μέρους του και ε, ε, ο πρόεδρος και άλλα μέρη της Επιτροπή ΣΥΝΤΑ, Κριστοβράου, Μαρία Μπάλντι, Τζόρτζ Κιούτας, και Μαρία Σάνκα. Σα συμμετείχαν από 29 Νοεμβρίου με 1η Δεκεμβρίου στη 23η Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση ε, στη Washington, το λεγόμενο TLD, τον Υπερατλαντικό Διάλογο και είχαμε, έγινε μια θαυμάσια συναδρίαση με την Κοινή Επιτροπή της, ε, του Κογκρέσου και ο Ντέβιτ Κάμπ προείδρευσε τη συνεδρίαση και ο πρόεδρος της υποεπιτροπής Κέβιν Μπρέιντι. 18 μέλη συμμετείχαν στην ε, Επιτροπή αυτή ε, και επίσης έγιναν και διμερείς συζητήσεις παραδειγματικές και για πρώτη φορά είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια άμεση συζήτηση για το πώς θα προωθήσουμε την, ε, το υπερατλαντικό εμπόριο τη συνεργασία μας λοιπά και να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και εκδηλώθηκε μια απόλυτη στήριξη σε αυτό το στόχο. Επίσης καλέσαμε εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου Κάναμε μια ξεχωριστή συναντήση με την πρέσβυρα Μίριαμ Σαπύρο, και μαζί με την, τον πρόεδρο, τον Κρίστιαν Έλερ, που είναι πρόεδρος της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, ε, συζητήσαμε και με τον Σύμβουλο Επισεμάτων Εθνικής Ασφαλείας και με εκπροσώπους ε, του Υπουργείου Οικονομικών για οικονομικά θέματα του υπερατλαντικού διαλόγου. Κύριε Κιούτας, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τίποτα να προσθέσω, ειδικά δεν θέλω, αλλά αφού έχω την ευκαιρία, ήθελα να πω ότι οι συζητήσεις που κάναμε ήταν εξαιρετικές και αυτό που έχει σημασία είναι η συμμετοχή των συναδέλφων μας από το Κογκρέσο το Αμερικανικό Κογκρέσο, η οποία ήταν πολύ άρισμη. Αυτό ήταν πολύ καλό για τις διαβουλεύσεις, για τις συζητήσεις και πραγματικά αυτές οι διαβουλεύσεις για τη νέα Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου έχουν λάβει μια καινούργια όθηση, έχει οριμάσει ο χρόνος και τα ενδιαφερόμενα μέλη υποσχέθηκαν να προχωρήσουν περαιτέρω έτσι ώστε σύντομα να έχουμε κάτι σημαντικό να ανακοινώσουμε στην Επιτροπή ο Προεδρεύων. Ναι, συμφωνούμε όλοι με αυτά που είπες. Πραγματικά θα εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία προόδου. Είναι μια καλή ευκαιρία για την Ευρώπη. Όσοι μείνετε μέχρι το τέλος αύριο, έχουμε μία πρόσκληση για ένα κοκτέιλ μετά από το τέλος της πρωινής συνεδρίασης στις 12.30 έξω από την αίθουσά μας. Όλοι είναι καλεσμένοι, το προσωπικό και τακτικά τα προσκεκλημένοι τα μέλη του προσωπικού και επίσης αύριο στο Paul Henry's Park 3Γ 3CO05 θα γίνει η συνεδρίαση. also uh, Η συνεδρίαση μας. Ο Ανδρέ θα φύγει από την γραμματεία μας μετά από τρία χρόνια επιτυχούς συνεργασίας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις μελλοντικές σας δραστηριότητες στην Ήτρε. Ήτρε, εν πάση περιπτώσει, εκεί. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό σε εμά. Πάντως ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα σου επιτροπή. Τέσσερα. Η πρόοδος των τριμερών διαπραγματεύσεων. Στις 5 Δεκεμβρίου ο πρώτος εισαγωγικός τριμερής διάλογος ε, έγινε για την ε, πρόταση του κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συμβουλίου που τροποποιεί την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ε, διαδικασία υιοθέτησης ορισμένων μέτρων. Η συγγήτριά μας δεν είναι εδώ τώρα. Μήπως ε, θέλει κανείς, έχει τίποτα να σχολιάσει για το 4. Ε, όσον αφορά τις, ε, τελωνια, την τελειωνιακή εφαρμογή των πνευματικών δικαιωμάτων, η, ο Ιώσεφ Αντρέα Μπέρα είναι συγητής της ΣΥΝΤΑ ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες, διευθύνωση επιτροπή ΙΜΚΟ και οι διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν αυτή την εβδομάδα. Από την κυρία Ανδρέα Μπέρερ, η οποία και αυτή λείπει. Το δεύτερο είναι ε, μηχανισμοί εταιρικής συνεργασίας, μηχανισμοί για την εδραίωση μιας συνεργασίας με τρίτες χώρες. Η συγητής, α, η συγγήτρια είναι η κυρία Ντρέτσκα και αυτή λείπει σήμερα. Ε, δεν, δεν τα πάμε και πολύ καλά, όλοι λείπουν φαίνεται. Τέλος πάντων, προχωρούμε στο 5. Δραστηριότητες, εποπτικές ομάδες, ανταλλαγή απόψεων. Κεντρική Ασία. Ε, συνεδρίαση έγινε στις 7 ε, ενδεκάτου με τα μέλη της ομάδας αυτής. Ε, έχετε τίποτα να προσθέσετε? Ναι, για το 5. Είχαμε μία συνεδρίαση, μία συνάντηση στις 7 Νοεμβρίου. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση της Υποπτικής Ομάδας για την Κεντρική Ασία και μας ενημέρωσε η Κομισιόν για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις και με το Καζακστάν και γενικά μας έδωσε τη συνολική εικόνα της περιοχής, τι γίνεται. Επίσης παρέστησαν και συνάδελφοι που είχαν επισκεφθεί την περιοχή πρόσφατα. Συζητήσαμε οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις για το PCA. Τα τελευταία νέα είναι ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα νέα, δεν έχει επιτευχθεί καμιά καινούρια πρόοδος σε αυτές τις διαβουλεύσεις και παρόλο που έγινε μια συνάντηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής και του Καζακστάν μετά από τη δική μας συνεδρίωση της εποπτικής ομάδας στις 14 Ενδεκάτου. Αυτό έγινε επειδή το Καζακστάν εστιάζεται αυτή τη στιγμή στο να γίνει μέλος του ΠΟΕ και υπάρχουν ορισμένα επίμαχα θέματα όπως εξαγωγική, δασμή κλπ. Ε, επίσης συζητήσαμε και όλα τα άλλα θέματα που άπτονται της Κεντρικής Ασίας, όχι τόσο πολύ εμπορικά όσο ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα. Ήταν μια γενική συζήτηση, οι συνάδελφοί μας έθεσαν πολλά ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα και βεβαίως τις δυνατότητες ανάψυξης του εμπορίου και συγκρίναμε τις διαφορές μεταξύ των χωρών και επίσης ε, συζητήσαμε τι μπορεί να προκύψει από προτάσεις της Κομισιόν στο μέλλον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έτσι ένα ολοκληρωμένο όραμα για ή προσανατολισμός που θέλουμε να πάμε. Γίνονται διαβουλεύσεις, αλλά τίποτα πιο συγκεκριμένο δεν προβλέπεται παρά η ανάλυση της γενικής εικόνας, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό, σε αυτή τη συνάντηση και προβλέπουμε με χαρά την συνεδρίαση της επόμενης, ε, την επόμενη συνεδρία τη εποπτική Ομάδας. Υπάρχουν σχόλια, όχι από κανέναν. Μεξικό, ε, στην ε, επόμενη συνεδρίαση. Ε, δεύτερη συνεδρία τη εποπτική Ομάδας. Καλέσαμε τον πρέσβη του Μεξικού στο Βέλγιο. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Αφορούσε την σημερινή κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού κατόπιν της ε, ε αλλαγής κυβέρνησης μετά τις τελευταίες εκλογές. Ε, το Μεξικό έχει καινούριο πρόεδρο. Ανέλαβε τα καθήκοντα του στο τέλος Νοεμβρίου. Οι Μεξικάνοι θέλουν να αναβαθμιστεί η ε, Συμφωνία Ελεύθερου ε, Εμπορίου με το Μεξικό. Εν τω μεταξύ, ε, συζητούμε μια παρόμοια συμφωνία με το Καναδά, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε είναι σημαντικό και για το Μεξικό να μην χάσει το τρένο. Όλοι οι συνάλφοι που ήταν παρόντες θα συμφωνήσουν μαζί μου. Πέραν του εμπορίου συζητήσαμε και θέματα ναρκωτικών, εμποριόπλων και άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους συναδέλφους στο Κοινοβουλίου. Ίσως στην επόμενη συνεδρίαση της εποπτικής ομάδας θα ήταν σημαντικό να εντοπίσουμε εκ των προτέρων ένα συγκεκριμένο θέμα, γιατί σε μία ώρα είναι αδύνατο να συζητηθούν τα πάντα. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους που ήρθαν στην έδρα της Υποπτικής Ομάδας. Thank you, George. Ωραία. Θέλει κανείς το λόγο να σχολιάσει. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Ε, οι τρεις συγκεκριμένες χώρες, οι ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό, αποτελούν μια ομάδα και θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα, όχι μαζί, αλλά ε, παράλληλα προς μια συμφωνία. Οι ΗΠΑ, εισηγητής είναι ο κύριος ε, Μορέιρα, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Συναντήθηκαν και αυτοί στις 28 Νοεμβρίου. Καναδάς, Πίτερ Στάσνη δεν είναι εδώ. Ντάνιελ, έχεις το λόγο. Ναι, αγαπητέ Ρόμπερτ, ο Πίτερ Στάσνη μου ζήτησε να πω μερικά λόγια, γιατί έγινε μια συνεδρία υποπτική ομάδα με τον Καναδά. Ήταν παρούσα η Κομισιόν και ενημέρωσε για τι τρέχουσε διαπραγματεύσεις. Και δεν πιστεύω ότι αποκαλύπτω τίποτα καινούριο, αλλά υπάρχει η ελπίδα να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, οπότε θα μπορέσουμε να ξαζητήσουμε αυτό το θέμα ενδελεχώς στην Επιτροπή μας. Ωραία, και εγώ το ίδιο είχα ακούσει, πιθανώς μετά τα Χριστούγεννα. Καλά τα νέα. Μαγκρέπ κυρία Δεσάρνα, δεν είναι εδώ, Βιετνάμ, ο κ. Ζαροντήλ είναι ο μόνιμος ηγητής και αυτός μας ενημέρωσε ότι δεν είναι εδώ, δεν θα μπορέσει να ήρθει. Θα μας ενημερώσει όμως τον Ιανουάριο. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Ο Ντάνιελ θα μιλήσει, ο εκ όχι, του εισηγητή. Περνάμε στο σημείο 5. 8 βασικά. Το 8 Ε, μάλλον θα συζητήσουμε το θέμα των ανανεώσιμων. Ε, έκθεση INI. Ε, προβλέπεται γνωμοδότηση από την Επιτροπή μας. Γιάννη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι είναι ενδιαφέρον σημαντικό το θέμα. Ιδιαίτερος στη σημερινή συγκυρία η Επιτροπή μας ε, στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου υπέβαλε μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για το κινέζικο dumping στα φωτοβολταϊκά πάνελς διαπιστώνουμε ότι εδώ και πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη σε μια φιλόδοξη πολιτική, κλιματική, πολιτική και ε, περιβαλλοντική πολιτική κλπ. Ε, έθεσε ε, στόχους για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ταυτόχρονα ανέπτυξε και μια βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, πολύ καινοτόμα και ανταγωνιστική, ε, δημιουργήσε με αυτόν τον τρόπο εκατοντάδε χιλιάδε θέσει εργασία στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να πείσουμε τα θεσμικά μας όργανα να αναπτύξουμε μια πολιτική που θα βασίζεται και πάλι σε αυτά τα δύο σκέλη. Πρώτον, φιλόδοξη περιβαλλοντική στόχη και από την άλλη μεριά από ανταγωνιστική βιομηχανία που θα δημιουργεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα δημιουργεί επιχειρήσεις σε όλη την επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια θα δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Σε αυτή την γνωμοδότηση προφανώς θα ξαναδούμε το θέμα των ε, παράνομων εμπορικών πρακτικών, εμπνεόμενοι κυρίως από την Κίνα και θα πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε μια ε, ανταγωνιστική και βιώσιμη βιομηχανία στην Ευρώπη αν δεν μπορούμε να αμυνθούμε έναντι τέτοιων αθέμητων πρακτικών. Δεύτερο σημείο το οποίο θα αναφέρουμε είναι η διεθνής διάσταση, επιθετικά πλέον, για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θεωρούμε για παράδειγμα ότι ε, κατόπιν των, της ε, διαδικασίας της Βαρκελόνης ε, και κατόπιν των όσων έχουν λεχθεί στο πλαίσιο της, Ένωσης για την, ε, ναι, της Ευρωμεσογειακής Ένωσης υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Νότια Μεσόγειο. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στις χώρες της Νότιας Μεσογείου να ικανοποιήσουν, να καλύψουν ένα μεγάλο τμήμα των αναγκών τους και γνωρίζετε το Desert Tech, το περίφημο σχέδιο ανάπτυξη ε, ε, φωτοβολταϊκών στην έρημο. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα δίναμε καθαρή ενέργεια στον νότο της Ευρώπης και ενδεχομένως θα μπορούσαμε βέβαια να υποφεληθούμε και με πολλούς άλλους τρόπους. Τέλος, θα αναφέρουμε την βιωσιμότητα της ε, παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, είναι ένα στοιχείο καινοτόμο, είναι ένα στοιχείο ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας. Η τεχνολογική καινοτομία θα μπορέσει να βοηθήσει την Ευρώπη αν επιτρέψουμε όχι μόνο να κατοχυρώσουμε τις εφευρέσεις αλλά και ταυτόχρονα να επωφεληθούμε και βιομηχανικά εμπορικά από, από αυτή την καινοτομία. Τέλος, κάτι που είναι λίγο επίμαχο στο εσωτερικό τη Κομισιόν, είναι το θέμα των κρατικών προμηθειών. Από την δική μου πλευρά, εγώ προσωπικά, πιστεύω ότι υπάρχει ένα θέμα γεωγραφικής προτίμησης. Δεν είναι δυνατόν ε, να θεωρούμε ότι το σύνολο των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων στον κόσμο ε, προσπαθούν να εξισορροπήσουν το άνοιγμα των αγορών τους με υποστήριξη των τομέων που είναι κρίσιμοι για τις οικονομίες τους ε, και χρησιμοποιούν εργαλεία όπως η γεωγραφική προτίμηση, για παράδειγμα η Βόρειος Αμερική αλλά και αλλού και δεν είναι δυνατόν αυτοί να το κάνουν και εμείς στην Ευρώπη ε, να ε, η, ελευθερία των εμπορικών ανταλλαγών να αφορά μόνο άνοιγμα της πρόσβασης ε, των αγορών μας. Πέραν της ε, αμοιβαιότητας, για την οποία θα βρούμε μια λύση, θα πρέπει να θέσουμε το θέμα της συλλογικής γεωγραφικής προτίμησης στο πλαίσιο των κρατικών προμηθειών. Όταν αντιμετωπίζουμε όλοι οικονομικά προβλήματα δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε ένα τόσο σημαντικό εργαλείο ε, της εμπορικής μας πολιτικής ε, όταν ε, μιλάμε για το 19% του ΑΕΠ μας. Ε, ο χρόνος πιέζει γιατί εμείς θα πρέπει να ετοιμάσουμε τη γνωμοδότηση μέχρι να επιστρέψουμε μετά τις διακοπές. Θα συζητηθεί το Γενάρη και αν δεν κάνω λάθος θα τεθεί προσιοθέτηση από την Επιτροπή στις 20-21 Φεβρουαρίου. Οπότε τροπολογίες θα γίνουν δεκτές μέχρι 28 Ιανουαρίου και κατόπιν θα περάσει την Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Yeah, thank you, Um, yes, I actually agree with... Συμφωνώ με τα περισσότερα που όσα είπες, Γιάννεκ. Υπάρχουν σχόλια. Αν όχι, ευχαριστούμε κύριε Χάους που ήρθατε. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να κάνετε κάποιο σχόλιο πλευράς τη Κομισιόν. Ε, ε, για τα όσα είπατε μόλις τώρα, υπάρχει μια σημαντική εμπορική διάσταση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων. Πολλά πολλοί συντελεστέ ε, επηρεάζουν την ανάπτυξή του. Ε, η Κίνα και η σχέση μα, για παράδειγμα, είναι ένας τέτοιο παράγοντας, ένα συντελεστή. Ε, Αναφερθήκατε για το Desert Tech, το πρόγραμμα ανάπτυξη των ανανεώσιμων στην Βόρεια Αφρική. Η συνεισφορά σα στην υπογράμμιση των ωφελών που μπορεί να, των ωφελιών που μπορούν να προκύψουν από την εξωτερική μας πολιτική και την ε, πολιτική εξωτερικού εμπορίου θα είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμες. Γιάννεκ. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν που είναι παρούσα. Ευχαριστώ πολύ. Well, it's always good to wish the Commissioner happy... Πάντα καλό είναι να ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά στον Επιτροπή. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, νομίζω ότι έχουμε τις βασικές ημερομηνίε. 23-24 Ιανουαρίου θα εξετάσουμε την γνωμοδότηση. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων 17 και 18 Δεκεμβρίου, που είναι σήμερα δηλαδή. Εξέταση σχεδίου έκθεσης 23 και 24, προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών 26 Φεβρουαρίου, ως γνωστόν μέχρι τις 12. Έγκριση της γνωμοδότησης 20 και 21 Μαρτίου στην Επιτροπή. Μη, σύντομο το χρονοδιάγραμμα λοιπόν, αν υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ή αν υπάρχουν και ενστάσεις, καλό θα είναι να φροντίσετε να τις κάνετε. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 6. Εισαγωγέ ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντέ. Ο Πολ Μέρφυ είναι ο εισηγητή. Έχουμε λοιπόν μια πρόταση κανονισμού για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές. Ε, σκοπός είναι να ευθυγραμμίσουμε τον υφιστάμενο κανονισμό με την διαδικασία επιτροπολογίας που προκύπτει από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο Πολ. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, αυτός είναι ο στόχος του νέου κανονισμού όπως και με, τους, ε, με τα θέματα Omnibus ε, και πολλούς άλλους ε, άλλα θέματα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διαφοροποίηση που γίνεται μεταξύ πράξεων κατοξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αρκετά τεχνικό λοιπόν το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι μας δίνει και μια εξαιρετική ευκαιρία να εξετάσουμε τα ευρύτερα ζητήματα κυρίως ε, το θέμα της πείνας και του στο στον Μπαγκλαντές και να κάνουμε και κάποια σχόλια τουλάχιστον γενικής φύσεως. Κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι το ρύζι είναι περίπου το 75% της γεωργικής παραγωγής του Μπαγκλαντές. Το 70% της συνολικής ε, ε, διατροφής των κατοίκων του Μπαγκλαντές και είναι και μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ. Επομένως αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομίας της χώρας και παρά το γεγονός ότι γίνονται εξαγωγές ρυζιού είναι μια χώρα που έχει έλλειψη τροφίμων και είναι και μια χώρα που έχει μεγάλη διατροφική ανασφάλεια. 65 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προβλήματα για την έβρεση και το 1 τέταρτο βρίσκονται κάτω από το όριο της στόχιας. Επομένως είναι πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία και μας εντυπωσιάζει και η φύση της γεωργίας. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των πολύ μικρών ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 86% ε, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι κάτω του ενός στρέμματος, ενώ ένα 10% είναι μόλις τρία στρέμματα. Ε, είναι πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία λοιπόν για τη γεωργία στον Παγκλαντές και η εξαγωγή γιου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον ε, βοηθά στην αύξηση των εισοδημάτων από το ρύζι και στην ε, βιωσιμότητα των ε, εσοδιών ώστε να μπορέσει να υπάρχει επάρκεια. Θα πρέπει βέβαια προκειμένου να έχουμε επάρκεια να επεκτείνουμε την παραγωγή η οποία θα είναι αντίστοιχη με την αύξηση του πληθυσμού που προς το παρόν είναι μόνο 2% ετησίως. Τώρα το πώς μπορεί να γίνει, ε, δεδομένου ότι οι περισσότεροι είναι μικροί γεωργοί στη χώρα τους, θα πρέπει να μπορούν να βρουν τρόπο να εξασφαλίσουν και τα τρόφιμά τους και τη βιωσιμότητά τους και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται αύξηση στην άρδευση, χρειάζεται μεταρρύθμιση στα θέματα των γεών και επίσης μεταφορά τεχνογνωσίας από πιο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτά λοιπόν ως γενικά σχόλια για την κατάσταση του ρυζιού στον Μπαγκλαντέ. Όσον αφορά το ίδιο το θέμα τώρα, σε πολλές ε, ε, πτυχές μπορούμε να, ακούσουμε, να ακολουθήσουμε τα όσα έχουν γίνει με τα θέματα Omnibus και να ακολουθήσουμε τις ίδιες άγουσες για να αυξήσουμε την δυνατότητα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, τις οποίες προτείνουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχε τροπολογίες που κάναμε και στα θέματα Omnibus. Παραδείγματο χάρη στο άρθρο 4 παράγραφος 2 αντί να δίνεται εξουσία στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή των κατεξουσιοδότηση πράξεων θα πρέπει να δίνεται μόνο για πέντε χρόνια, ε, τα οποία θα παρατείνονται για άλλα πέντε χρόνια και ούτω καθεξής. Και αντιστοίχως, στο άρθρο 4 σημείο 5, στην περίπτωση που το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέλουν να έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να εξετάσουν ένα διάστημα, θα πρέπει να είναι τέσσερι μήνε αυτό το μεγαλύτερο διάστημα και όχι δύο μήνε. Και υπάρχουν και μια σειρά από άλλα στοιχεία αντίστοιχα ε, και έχω και κάποιε συγκεκριμένε ερωτήσεις προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα θέσω σήμερα ή να προκύψουν και από τις συζητήσεις αργότερα. Υπάρχει κάτι νέο το οποίο δεν υπήρχε στις προηγούμενες προτάσεις κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ελαιόλαδο. Η τελευταία φράση της αιτιολογικής σκέψης 4 που αναφέρεται στο άρθρο 1 ε, παράγραφος 3. Η τελευταία φράση χωρίς να εφαρμόζεται ο κανονισμός 182 του 2011, μας επιτρέπει να έχουμε μια παρέκκληση ε, για τις εκτελεστικές εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ερώτημά μου είναι κατά πόσον, γιατί θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη για εξαίρεση αφού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στους άλλους κανονισμούς που προτείνει και γιατί δεν επαρκεί ε, όταν καθαρίζεται το όριο των ποσοστώσεων, ε, που είναι 4.000 τόνοι, να μπορεί να δράσει απευθεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει αυτό το ποσοστό. Και στα άρθρα 7 και 8 του σχετικού κανονισμού 182 του 2011, το οποίο αναφέρεται στην άσκηση ελέγχου των κρατών μελών ε, στα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, γιατί λοιπόν, αφού αυτό μας καλύπτει, γιατί πρέπει να γίνει αυτή η εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανονισμό για να μπορούν να ανταποκριθούν ε, στις απαιτήσει. Υπάρχουν ωφέλη ε, στο τα πάντα εκτός από όπλα. Υπάρχει περίπτωση να ισχύει αυτό σε πραγματικούς όρους αν ε, το Μπαγκλαντές χάσει το, τα πάντα εκτός από όπλα και θα πρέπει ε, να βασίζονται σε κάτι το οποίο πρέπει να γίνει αλλά τελικώς δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Τέλος, να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για τη βοήθειά τους μέχρι τούδε και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζορ Κουτάς. Ευχαριστώ καταρχάς να εξηγήσω ότι εγώ δεν είμαι ο ηγητή από πλευρά τη ομάδας μου. Αντικαθιστώ τον Τζαν Λούκα και ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του γιατί δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα. Η άποψή του για τη συγκεκριμένη συζήτηση είναι η εξή η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στόχο έχει να ευθυγραμμίσει τον κανονισμό για τις ε, εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές ε, και να τον ευθυγραμμίσει στις αλλαγές που έγιναν με την εισαγωγή της συνθήκης της Λισαβόνας και κυρίως να ρυθμίσει τα θέματα κατεξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων που ρυθμίζονται στα άρθρα 290 και 292 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρόταση αυτή και υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για να βρούμε την κατάλληλη διαδικασία για να εγκρίνουμε τις πράξεις αυτές οι οποίες απορρέουν από τον κανονισμό. Ε, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν πράξεις κατεξουσιοδότηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καθορίζονται τα θέματα συμμετοχής ε, και να ρυθμιστεί το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας. Επίσης υπάρχουν κάποια διοικητικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των προτιμησιακών καθεστώτων, εισαγωγή, ε, την περίοδο ισχύω ε, της χώρας καταγωγής, ε, την περίοδο ισχύω της άδειας εισαγωγής, όλα αυτά θα πρέπει να ρυθμίζονται με εκτελεστικέ πράξεις. Η άποψή του αυτή τη στιγμή είναι ότι θα ήθελε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή συνοχή με τον κανονισμό Omnibus, και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στη διάταξη η οποία ήδη εγκρίθηκε στο Όμνιμπος και την υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εκχώρηση των αρμοδιοτήτων ε, μόνο για τα πέντε χρόνια μετά από την έγκριση του συγκεκριμένου κανονισμού και την, ε, ε, τις διαβουλεύσεις για τις εξαγωγές. Επίσης, ο Τζαν Λούκα έχει θετική στάση ως προς την ε, έκθεση και είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί και με τους και κοιόδης συγητέ και τον εισηγητή για το θέμα αυτό. Η Φραντσέσκα Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις γενικές σας παρατηρήσεις και για τον Μπαγκλαντές και ιδίως ε, τα προβλήματα της γεωργίας που αντιμετωπίζει λόγω της αλλαγής του κλίματος ε, με βρίσκουν σύμφωνα τα όσα είπες. Έχω κάποιες ερωτήσεις τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάποια θέματα τα έχουμε ήδη θίξει. Την αναστολή των μέτρων όταν εξαντλούνται ποσοστώσεις. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ε, να δράει η ίδια χωρίς βοήθεια της Επιτροπής Επιτροπολογίας. Ε, σκοπεύει να αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς ε, την Επιτροπολογία ε, όπως συνέβαινε στον κανονισμό 3490-90. 91-90. Πρώτη ερώτηση αυτή και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ασκούνται πράξεις κατεξουσιοδότηση για να καθορίζονται τα θέματα των εισαγωγών μέσω μιας διαδικασίας ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό το lodging of security, τι ακριβώς εννοείται με αυτό που αναφέρεται εδώ. Και επίσης το να ρυθμίζετε το θέμα της ασφάλειας και να εξαρτάται από αυτό το προτιμησιακό καθεστώς τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση με τις εγγυήσεις που ζητάτε. Να ρωτήσω επίσης γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει συμπεριλάβει το κανονισμό αυτό σε όλο τη δέσμη μέτρων του Omnibus, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ομοιομορφία στην νομοθεσία. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ Φραντσέσκα. Υπάρχει εκπρόσωπος εδώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι συνεκτικό με τα όλα θέματα όμνιμπους, αυτό είναι δεδομένο. Δεύτερον, ρωτήσατε γιατί δεν χρειάζεται τη συνδρομή επιτροπής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον εξής λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει απλώς ένα μαθηματικό υπολογισμό για να δει κατά πόσον έχουν ε, φτάσει αυτά τα ανώτατα όρια. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ευελιξίας εδώ και δεν υπάρχει κανένας όλοχος, ε, καμία ανάγκη ελέγχου από τα κράτη-μέλη. Να σας παραπέμψω στην αιτιολογική ε, σκέψη 6 το έχω μόνο στα γαλλικά το κείμενο, αλλά στον κανονισμό αυτό, τον 182, α, το έχω και στα αγγλικά εδώ, λέγεται ότι εφαρμόζεται στις βασικές πράξεις που απαιτούν τον έλεγχο των κρατών μελών. Δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται έλεγχος γιατί απλώς θα εφαρμόσουμε ένα μαθηματικό τύπο και επίσης δεν υπάρχει ανάγκη να διασφαλίσουμε ομοιόμορφε συνθήκε εφαρμογέ, Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 1. Πρόκειται απλώ για ένα μηχανικό υπολογισμό. Μόλις φτάσουμε σε αυτά τα ανώτατα όρια, γίνεται ένας απλός μαθηματικός υπολογισμό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει απόφαση. θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει και αν πρόκειται για νομική πράξη αυτή την περίπτωση. Είναι απλώς μια συνηθισμένη πράξη. Και γιατί δεν το έχουμε σωματίσει αυτό στα υπόλοιπα θέματα όμνιμπους, δυστυχώς δεν μπορώ να σας απαντήσω, θα προσπαθήσω να διαπιστώσω γιατί έγινε αυτό. Αυτό λοιπόν έχω να σας απαντήσω. Δεύτερον, ρωτήσατε κατά πόσον ο κανονισμός ισχύει μόνο όταν δεν εφαρμόζεται τα πάντα εκτός από όπλα. Έχετε δίκιο, όντως ο κανονισμός αυτός δεν εφαρμόζεται καθόλου, διότι, διότι ισχύει το everything but arms. Και τρίτον, το θέμα της εγγύησης. Αυτό είναι ένα τεχνικό μέτρο το οποίο συχνά επιβάλλεται στη διαχείριση των ποσοστώσεων, ζητείται από τους εισαγωγείς να καταθέσουν μια εγγύηση για να διασφαλίσουμε ότι είναι σοβαροί και ότι δεν ζητούν απλώς να κάνουν μια εισαγωγή και μετά να κερδοσκοπήσουν να κάνουν εμπορία. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι εισαγωγεί απλώς θέλουν να κάνουν εισαγωγή και γι' αυτό ακριβώς τους ζητείται να καταθέσουν εγγύηση. Αυτό είναι ο λόγο. Απάντησα όλες σα τις ερωτήσεις. Ναι, σύντομα. Ευχαριστώ την Κομισιόν και τους σκιώδεις εισηγητές για τις απαντήσεις τους και συμφωνώ με όλα αυτά τα σημεία που εισήγησαν πρέπει να συμφωνεί με τις ε, προτάσεις του Omnibus ασφαλώς και μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτές τις προτάσεις που περιλαμβάνουν την παραπομπή ε, στους εμπειρογνώμενους, δηλαδή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα πρέπει να βρούμε και να εξετάσουμε εάν αυτή η διαδικασία είναι η σωστή για να μπορέσει να υιοθετήσει εκτελεστικές ε, πράξεις ή κομισιόν χωρίς την ε, Σύνδρομη Επιτροπής. Από την πλευρά μου λοιπόν θα εξετάσω αν μπορούμε να κάνουμε παρόμοιους κανονισμούς χωρίς αυτό και αν αυτό είναι καλύτερη μέθοδος παρά να αναστείλουμε την ισχύ κανονισμών. Ε, καταλαβαίνω το επιχείρημα ότι ασφαλώς ε, βάση του άρθρου 1.3 μιλάτε για μια ποσότητα 4.000 τόνων και όλη αυτή η ανάλυση ε, παρουσιάζεται καλύτερα στο εκτιμώντας 4 αιτιολογική σκέψη 4, γιατί λέει ότι αν γίνει αναστολή των προτιμησιακών ρυθμίσεων κτλ, η Κομισιόν θα πρέπει να, να δοθεί δυνατότητα στην Κομισιόν να υιοθετήσει εκτελεστικές πράξεις χωρίς ε, την εφαρμογή του κανονισμού. Ε, Πρέπει λοιπόν να δούμε και την πλευρά των πολιτικών αποφάσεων ε, και γι' αυτό προτείνω να καθυστερήσουμε την προθεσμία για την έκθεση αυτή έτσι ώστε να μπορέσουμε να μελετήσουμε ακριβώς τις θέσεις των ενδιαφερομένων και της Κομισιόν και να δούμε ότι πραγματικά συνάδουν με το πακέτο Omnibus. Πρόεδρος, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή, την Κομισιόν, αν θέλει να δευτερολογήσει. Ρώτησα και τη Γραμματεία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αναστολής. Θα αναστείλουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Αν συμφωνούν οι σκιώδεις εισηγητές, κανένα πρόβλημα. Η Επιτροπή δεν έχει τίποτα να προσθέσει. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε Πολ. Και προχωράμε το 7 αποστολή στην Ιρλανδία. Όπως ξέρετε, μια πολύ άρισμη ε, αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Δουβλίνο στις 6 Δεκεμβρίου εν ώψη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ήταν ο David Μάρτι, George Κιούτας, Μπέρνατ Λάγκε, Κάθριν Μπίρντερ και ο Πολ Μέρφυ και βεβαίως ο Πρόεδρος. Θα διαβάσω τη σύντομη ε, ανασκόπηση της επίσκεψης αυτής εκ μέρους του Πρόεδρου. Λέει λοιπόν ότι κατά τη σύντομη επίσκεψή μας συναντήσαμε τον Υπουργό Επιτρο... ε, Επικρατείας τον κύριο Σέρλικ, επίσης εκπροσώπους της Ιρλανδικής Επιτροπής Εμπορίου, μέλη ε, του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Έχει μια παράξενη ονομασία το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο που δεν ξέρω πώς να την πω. Τέλος πάντων ε, συναντήσαμε και βουλευτές, ε, είχαμε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και με την Επιτροπή Εμπορικών Συναλλαγών, επίσης διάφορους εκπροσώπους ε, από την Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών και Εργοδοτών, από την Ιρλανδική ΓΕΣΕΕ και την Ένωση Εξαγωγέων και επίσης επισκεφθήκαμε και τα γραφεία της Google την επόμενη μέρα είχα μια διμερή συνάντηση με τον ε, Υπουργό Μπρούτον, ο οποίος είναι υπουργό Εργασίας και ε, συζητήσαμε βεβαίως και με τον αρμόδιο Υπουργό την κοινή εμπορική πολιτική. δεν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν επισκέφτηκαν το εργοστάσιο της Γκίνες. Δεδομένου ότι η Γκίνες είναι ένα τόσο αντιπροσωπευτικό Ιρλανδικό προϊόν. David, τι έχεις να πεις. Ευχαριστώ Ρόμπερτ, δυστυχώς δεν διαμόρφωσα εγώ το πρόγραμμα. Ε, να προσθέσω σύντομα, αυτό που προέκυψε από την συνάντηση είναι πόσο σημαντικό είναι το, οι εμπορικές συναλλαγές για την Ιλλανδία ως χώρα και βεβαίως το θέμα πόσο σημασία έχει για την επερχόμενη Προεδρία. Είχαμε πολλές ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων για τις εμπορικές συναλλαγές και ε, με χαροποίησε, με ικανοποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλοι οι εκπρόσωποι, όλοι οι συνομιλητές μας ήταν πολύ καλά ενημερωμένοι για τα επίκαιρα θέματα. Η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει τις διαβουλεύσεις με την Αμερικανική πλευρά για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου δεν ξέρω αν αυτές οι συνομιλίες, οι διαβουλεύσεις ολοκληρωθούν υπό την Ιρλανδική Προεδρία, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να προωθήσουν το θέμα αυτό και να προωθήσουν και άλλους φακέλους όπως το Omnibus και επίσης το ντοσιέ της πρόσβασης στις αγορές. Ε, τα θέματα αυτά θα έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας τους. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και δραστήρια Προεδρία. Σε ευχαριστούμε, David. Ε, άλλα σχόλια, παρακαλώ ο Βίλιαμ. Διάβασα αυτήν την έκθεση με κάποια δυσπιστία ή ε, κάποια περίεργη αντίδραση, διότι δείχνει τι ε, μεγαλειώδεις εξελίξεις ή τι μεγαλειώδης κόσμος ε, υπάρχει στην Ιρλανδία και τι καλά που πάνε τα πράγματα μεταξύ Ιρλανδίας και Ευρώπη. Η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια τεράστια κρίση και ε, συναντήθηκε η Επιτροπή με την Ένωση Εργοδοτών, με την Ένωση Εξαγωγέων, με την Ιρλανδική ΓΕΣΕ, τα συνδικάτα κλπ ε, και κάποια αναφορά γίνεται ότι η Ιρλανδία τώρα επικύρωσε ένα πάρα πολύ αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας. Τώρα το θέμα όμως είναι τι γίνεται με την άποψη των Ιρλανδών ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας από αυτούς ε, δεν έχει άποψη για το αν θέλουν να είναι εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγχουν ε, τα συναλλαγμά τους από θέματα τη συναλλαγματική τους ισοτιμία, τα οικονομικά τους, αν θέλουν, να είναι δηλαδή αφεντικά του αυτού τους ή αν θέλουν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στο ζουλομανδία του ευρώ. Ε, κανένας δεν είπε την άποψή του. Εδώ έχουμε ένα ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο και κανένας δεν τον βλέπει. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τις απόψεις των ε, Ιρλανδών, της Ιρλανδικής Ένωσης εξαγωγέων. Πώς πιστεύουν ότι θα προωθήσουν τις εξαγωγές τους εάν τα δεδομένα της Ιρλανδικής οικονομίας είναι υπερβολικά υψηλά, υπερβολικά χαμηλά ή ακριβώς όπως πρέπει. Κάποια γνώμη δεν θα πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν εξαγωγέ. Και το βρίσκω πολύ παράδοξο ότι δεν διαπιστώνω καμία τέτοια αντίδραση εδώ μέσα, καμία τέτοια αναφορά. Ε, ε επίσης, ο Ιρλανδός εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ, των συνδικάτων, των συνομοσπονδιών, ε, δεν 12 ώρες συναντήσεων και καμία άποψη δεν εκφράστηκε. Ο συνάδελφός μας, Μέρφυ, έχει πει πάρα πολλές φορές τι δυστυχία, τι μιζέρια έχει δημιουργήσει αυτή η κατάσταση οικονομική της Ευρώπης στην Ιρλανδία, τις τεράστιες περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, στις δημόσιες δαπάνες, ανεργία και γενικά δυστυχία. Αυτή η αρνητική πλευρά δεν εφήγει καθόλου. Μήπως θα μπορούσε ο κύριος Μέρφυ να διαθέσει ένα λεπτάκι να μας φωτίσει ή τουλάχιστον να φωτίσει εμένα για το τι γίνεται. Σε ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Σε ευχαριστώ, ο Βίλιαμ. Από ό,τι κατάλαβα, η ομάδα σου συμμετείχε σε αυτή την αποστολή, μήπω. Θα μπορούσε και η Επιτροπή Οικονομικών Οίκων ήταν ε, επίση ε, στην Ιρλανδία την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Βίλιαμ, επί διαδικουστικού. Κύριε Πρόεδρε, είσαστε ένα πάρα πολύ ευγενή και εγωιτευτικό άνθρωπο και σα σέβομαι ιδιαίτερα. Όμω, ε, δεδομένου ότι εγώ είμαι μέλος εδώ και τρία χρόνια, τα μέλη της, της δικιάς μου ομάδας έχουν εντολή να μη συμμετέχουν στις αντιπροσωπείες. Α, ναι, λέει ο πρόεδρος που είναι 13 χρόνια στο σώμα. Ίσως είναι παραείμαι εδώ τόσα χρόνια. Ο Ντέιβιντ ε, κάτι θετικό θα προκύψει και από το να μην ταξιδεύει κανείς. Τουλάχιστον θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ντέιβιντ, λοιπόν, ε, εγώ είχα καλέσει τον κύριο Πολ Σουίνι πριν από τρία χρόνια ε, στο Εδιμβούργο, όχι το 2007, για να μας μιλήσει για την οικονομική κρίση στην οποία βρισκόμεθα τότε και είμαστε και τώρα. Και βεβαίως ε, κατηγορήθηκαν οι τράπεζες, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και επίσης κατηγορήθηκε ως βασική ένοχη οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου το Υπουργείο Οικονομικών επέτρεψε την πάρα πολύ εύκολη δανειοδότηση και πολύ χαλαρή χρηματοδοτική πολιτική. Είχαμε εκφράσει λοιπόν ε, τεράστιες ανησυχίες για το πρόγραμμα αυτό λιτότητας και την ανικανότητα της Ιρλανδίας να το αντιμετωπίσει και είχαμε ζητήσει να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας προς την Ιρλανδία. Αλλά θα ήταν μια πραγματική καταστροφή, όχι μόνο για την Ανωμένο Βασίλειο και για την Ιρλανδία, να αποσυρθεί, να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό θα σήμαινε και ένα τέλος της εξαγωγής και καταστροφή γενικώ. Δεν, δε δέχομαι το δόλωμα, λέει το μέλος που του δόθηκε ο λόγος. Ο Πρόεδρος, θέμα 8. Προσωρινή αναστολή τη συμμετοχή του Μιανμάρ στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. Πρώτη συζήτηση για την ε, ε, πρόταση της ε, αναστολής συμμετοχή της Μιανμάρ στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. Η συμμετοχή αυτή είχε ανασταλεί προσωρινά το 1998 εξαιτία. Ε, του, της εξαναστικής εργασίας που ε, χαρακτηρίζει την Μιανμάρ. Ε, από το 2011 η Μιανμάρ ξεκίνησε όμως ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ε, κάτι που οδήγησε σε σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την ε, ικανοποίηση των προτάσεων του παγκόσμιου των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Σήμερα θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Κάρι τα πει όλα, ειδικό σύμβουλο του Γενικού Διευθυντή της Παγκόσμιας Οργάνωσης ε, Εργασίας. Καλωσορίζω τον, τον κύριο Τσέφολ της ITUC. Κύριε Ταπιόλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας εξηγήσω ποια είναι η κατάσταση από πλευράς ILO. Έχουμε σημαντικές, ε, ε, ε σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την, τη Σύμβαση 29 και τη Σύμβαση 87. Ε, όλα αυτά έχουν αλλάξει το πλαίσιο στο οποίο κινείται η Διεθνής Οργάνωση Εργασία ε, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Μιανμάρ. Φέτος ελήφθησαν ε, αρκετές αποφάσεις. Ε, συζητήσαμε στην αντίστοιχη επιτροπή ε, την εφαρμογή των συμβάσεων ε, ιδιαίτερα σε αφορά την καταναγκαστική εργασία. Έγινε συζήτηση με την κυβέρνηση. Η Επιτροπή Ευρωμόνων του ILO τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο προέβη σε μια αξιολόγηση της κατάστασης. Η έκθεση αυτή όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Πριν από 10 μέρες δημοσιεύθηκε το πρώτο, η πρώτη εκδοχή της. Ε, τον Μάρτιο θα δημοσιευθεί η τελική, τελική της μορφή. Συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας αναφέρω το, τίποτα από το περιεχόμενό της. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, νομίζω ότι η Επιτροπή προνομών συμφωνεί με αυτά που λέω. Ε, σε ό,τι αφορά το ψήφισμα της διάσκεψης, η τους ε, περιορισμού σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την κυβέρνηση της Μιανμάρ. Αυτοί οι περιορισμοί είχαν καθοριστεί από παλιότερο ψήφισμα του 1999, ε, δεδομένου ότι η Μιανμάρ δεν συμμορφωνόταν με τις συστάσεις της ε, Ερευνητικής Επιτροπής. Η άρση των περιορισμών ε, επαναχορηγεί το πλήρες καθεστώς συμμετοχής της Μιανμάρ. Το, σε ένα από τα ψηφίσματα του 2000 υπήρχε μία παράγραφος την οποία πλέον αναστήλαμε μέχρι ότου ξανασυζητηθεί την επόμενη, τον επόμενο Ιούνιο. Είναι αυτή που καλεί τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν τη σχέση με τη Μιανμάρ συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών σχέσεων. Η διάσκεψη θα αναθεωρήσει αυτή την παράγραφο τον Ιούνιο του 2013. Ε, οπότε το Μάρτιο του 2013 όταν θα είναι έτοιμη η έκθεση ε, θα ε, μας δοθεί ευκαιρία να έχουμε και υλικό προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτή την αναθεώρηση. Πάντως το ψήφισμα του 2000 έχει ανασταλεί, δεν ισχύει πλέον τρεις από τις πέντε παραγράφους του ψηφίσματος που είχε ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΑΕΛΟ έπαψαν να ισχύουν. Μία από αυτές θα την δει το, ε, ε, ε το ε, τελεστικό όργανο. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι ε, μια ε, ελάχιστη στάση σόφρων. στάση καλούνται τα κρατημέλη και οι διεθνείς οργανώσεις να χορηγήσουν τις κατάλληλες οικονομικές, τα κατάλληλα οικονομικά κονδύλια, τα κατάλληλα κονδύλια μάλλον, για να βοηθηθεί η Μιανμάρ να καταργήσει την καταναστική εργασία μέχρι το 2015 και έχουμε ήδη ένα ε, σχέδιο, ένα project για την ελευθερία του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε. μάλιστα, ε, ε, κατευθείαν πήγαμε στη Μιανμάρ για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή. Η Μιανμάρ το Φεβράριο του 2012 υιοθέτησε ένα ε, νόμο ε, που τιμωρεί την καταναγκαστική εργασία. Ε, υπάρχουν και όμως και άλλες δράσεις, ευαισθητοποίησεις και στους πολίτες και στους στρατιωτικούς. Υπάρχει ένας πλέον μηχανισμός προσφυγής. Ήδη από το 2007 υπήρχε κάποιος ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί. Η εφαρμογή της ε, καταναλωτικής έχει μειωθεί, παρόλο ότι όμως υπάρχουν ακόμα πολλές καταγγελίες. Η κυβέρνηση εξακολουθεί ε, να κάνει μεταρρυθμίσεις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές ε, και έχουμε μια περίοδο μεταπολίτευσης μετά από πολλές δεκαετίες δικτατορικού καθεστώτος. Πρόκειται για μια σημαντική δέσμευση από πλευράς της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ε, δράσης κατά της ε, καταναγκαστικής εργασίας. Ε, σε υψηλότατο επίπεδο καταδικάζεται η καταναγκαστική εργασία, ιδιαίτερα αυτή από πλευράς του στρατού και, και ο, ο Πρωθυπουργός της Μιανμάρ έχει αναλάβει προσωπική δέσμευση να καταργήσει πλήρως την καταναγκαστική εργασία, κάτι το οποίο ζητούσε ο εδώ και πολύ καιρό. Η σημερινή κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι ε, έχει ως εξής. Η υιοθέτηση αυτού του νόμου εναντίον της καταναγκαστικής εργασίας ε, το Φεβρουάριο του 2012 είναι ένα ικανοποιητικό βήμα, ένα ικανοποιητικό μέτρο. Ιδιαίτερα ε, δεδομένου ότι συμπληρώθηκε από μια πρόσθετη τροπολογία που, για κάτι που είχε ξεχαστεί. Ε, απομένει να αναθεωρηθεί και το Σύνταγμα ε, σε ό,τι αφορά την ε, πτυχή των καθηκόντων των πολιτών σε θέματα κρατικού συμφέροντος, δημοσίου συμφέροντος. Ελπίζουμε ότι μεταξύ δεν θα τύχει κατάχρηση αυτή η ρήτρα του συντάγματος. Ήδη ο νόμος του Μαρτίου 2012 έλυσε το θέμα αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν ιδιαίτερα επίγοντα θέματα σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση καινούργια νομοθεσία με την εξαίρεση της ανάγκης ε, μεταρρύθμιση του συντάγματο. Η έμφαση θα δοθεί στην τεχνική συνεργασία από εδώ και πέρα ε, και, στο πλαίσιο, και παρουσιάστηκε στους δωρητές ένα πρόγραμμα πλαίσιο με τρεις βασικούς στόχους. Πρώτον, ε, καταναγκαστική εργασία. Σήμερα μάλιστα ήμουν σε επαφή με, τα, με το γραφείο μας στη Γιάνγκον και από εκεί μας αναφέρουν ότι το πρόγραμμα ε, εξελίσσεται. Ε, ένα άλλο σημείο είναι η ελευθερία του ε, συνεταιρίζεστε και η πρόθεση του κοινωνικού διαλόγου σύμφωνα με την Σύμβαση 87 περί του του συνεταιρίζεστε και ένα τρίτο στοιχείο του πρόγραμματος πλησίου είναι ε, ένα πρόγραμμα ε, αξιοπρεπούς εργασία. Κάτι δηλαδή θα είναι πιο γενικό, θα περιλαμβάνει ε, στοιχεία κοινωνικά και εργατικά. Να σας πω δύο λόγια για ένα θέμα από το οποίο είναι ανοιχτό και για το ψήφισμα που υιοθετήθηκε από τη διάσκεψη τον περασμένο Ιούνιο. Ζήτησε από τον ILO τον Νοέμβριο να υποβάλει έκθεση για την κοινή στρατηγική, την λειτουργία της καινούργιας εργασιακής εργατικής νομοθεσίας και τις ε, ε των ε, εξωτερικών, άμεσων ε, εξωτερικών επενδύσεων στις ε, εργασιακές συνθήκες. είναι αυτή η παράδοση η οποία θα ξανασυζητηθεί τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά τις ξένες άμεσες επενδύσεις, ε, είπαμε ε, στην έκθεσή μας ότι υφίσταται ε, ένα νόμος πλαίσιο για αυτές τις επενδύσεις στο Κοινοβούλιο. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, αλλά ελάχιστοι ξένοι επενδυτές έχουν ακόμα έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Ε, ιδιαίτερα για τον ε, τουρισμό, την ε, οικοδομή και τις δημόσιες υπηρεσίες. Εταιρική κοινωνική ευθύνη έχουν, έχει, έχουν αληθεί κάποιες δεσμεύσεις από πλευράς των επιχειρηματιών και πάνω από 100 εταιρείες έχουν υπογράψει τη σύμβαση. Έχουμε ε, συζητήσει με την κυβέρνηση Μιανμάρ, με επενδυτές και με προσώπους διαφόρων ε, άλλων κυβερνήσεων ε, για την εφαρμογή μοντέλων βέλτιστων πρακτικών, εθελοντικής συμμετοχής κλπ. Θα συνεχίσουμε να υποβάλουμε εκθέσεις στο διοικητικό όργανο, στο διευθυντικό όργανο συγγνώμη, του ILO. Ε, δύο λόγια τώρα για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Παρόλο ότι οι κυρώσεις δεν επιβλήθηκαν για την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, αλλά για την καταναστική εργασία. Παρ' όλα αυτά, ε, έγινε πρόταση για ε, τη χρήση του άρθρου 26 ε, της 87. Ε, Το άρθρο 26 ε, είναι το άρθρο το οποίο προβλέπει την δημιουργία μιας, ε, τη σύσταση μιας ερευνητικής επιτροπής. Ε, το διευθυντικό όργανο αποφάσισε όμως να μην αναλυφθεί η δράση με βάση αυτό το άρθρο. Αντιθέτως, το ILO να συνεχίσει την στενή συνασία με την κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά η Σύμβαση 87. Υπάρχει ένας καινούριο νόμος για τις εργαστικές, εργασιακές ενώσεις. Ε, βοηθούμε την ε, κυβέρνηση, την, ε, ε δίνουμε συμβουλές και έχουμε 264 εργασιακές ενώσεις, μία συνομοσπονδία και 12 ενώσεις εργοδοτών. Ε, ο πρόσωπος ITUC μπορεί να μας πει περισσότερα πράγματα γι' αυτά. Υπάρχει μια, ένας καινούριος νόμος για τη ρύθμιση, επίλυση εργατικών διαφορών. Είναι σημαντικός γιατί κατήργησε ένα παλιό νόμο του 1929. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ε, είχε ζητήσει την κατάργησή του στο παρελθόν. Ε, υπήρχε και ένα διάταγμα του 1988 για την ε, το, το, ε, παράνομο συνέρχεσθε, ε, κάτι που επίσης καταργήθηκε. Ο επικεφαλής των συνδικαλιστικών Ανώσεων της Μπούρμα επέστρεψε στη Γιάνγκόνα τον Οκτώβρη μέσω μιας διαδικασίας που, στην οποία συμμετείχε και ο ILO Ε, η κυβέρνηση έδωσε εγγύησεις σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του να ε, εργαστεί και ότι δεν θα του επιβληθούν κυρώσεις. Η ITUC έλαβε άδεια, <clears throat> έγκριση, να ανοίξει γραφεία και την περασμένη εβδομάδα ε, έλαβε χώρα ένα σεμινάριο κατάρτισης για συνδικαλιστές. Ήρθαμε σε επαφή με πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κύριε Πρόεδρε, αυτό ήταν μια σύνοψη της κατάστασης. Όπως σας είπα, δεν μπορώ να σας ε, αναφέρω αυτό λεξί ε, ε, κομμάτια της έκθεσης, ε, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Πλην όμως, ό,τι σας είπα, ευθυγραμμίζεται με τα απορίσματά της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φώτς από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο σήμερα Είμαι νομικό σύμβουλο ε, σε θέματα Ασία ε, για τη Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και ασχολούμαι με τα θέματα αυτά εδώ και κάποια χρόνια. Θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Καταρχά ε, για να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο συνάδελφο ο κύριος Ταπιόλα για αρκετά από τα θέματα τα οποία έφυξε στην παρουσίασή του. Ε, λίγο πολύ λοιπόν εγώ απλώς θα τονίσω περαιτέρω κάποια σημεία και θα σταθώ λίγο πιο συγκεκριμένα ε, στην άποψη ε, της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας ε, Συνδικάτων και στο τι φρονεί ότι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει την κατάσταση. Καταρχάς, για το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας, προφανώς η συστηματική χρήση καταναγκαστικής εργασίας ήταν αυτό το οποίο οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει το προτιμησιακό καθεστώς στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για τη Μιανμάρ. Έγινε μια έρευνα από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ε, και έγιναν και κάποιες συστάσεις. Ε, μία σύσταση ήταν να αλλάξει η νομοθεσία. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τέλος στην καταναγκαστική εργασία και επίσης να εφαρμοστούν και κυρώσεις ποινικού ε, δικαίου. Όσον αφορά τώρα την εξάλληψη της καταναγκαστικής εργασίας, όπως αναφέρθηκε υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με σκοπό να σταματήσει η καταναγκαστική εργασία μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, 31 Δεκεμβρίου, αλλά εξακολουθούμε μέχρι σήμερα να λαμβάνουμε καταγγελίες για καταναγκαστική εργασία, ε, την οποία επιβάλλει ο στρατός σε αρκετές περιοχές ε, ε, στη Μιανμάρ σε αρκετές ε, ε, περιοχές και αυτό φυσικά ε, γίνονται για πολλούς από τους σκοπούς που ακούσαμε, για υποδομές για το στρατό, δικά δίκτυα και ούτω καθεξής. Πιστεύουμε ότι υπήρχε μείωση στην άσκηση καταναγκαστικής εργασίας, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τη Βυρμανία. Κατόπιν, μια τρίτη σύσταση από την Ερευνητική Επιτροπή ήταν να εφαρμοστούν ποινικέ κυρώσει και από ό,τι βλέπουμε από τι πιο πρόσφατες εκθέσεις της Διεθνούς παρά το γεγονός ότι στο στρατό υπήρξαν κάποιες τιμωρίες, διοικητικές όμως κυρίως κυρώσεις, αναστολές, μειώσεις στους μισθούς κλπ. Μόνο τέσσερις στρατιωτικοί ε, φυλακίστηκαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από το 1998 και τούδε. Επομένως υπάρχει ατιμερησία και εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Μόνο τέσσερα άτομα φυλακίστηκαν για καταναγκαστική εργασία. Όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουμε δει πολύ ουσιαστικές βελτιώσεις. Ε, υπάρχουν πλέον συνδικάτα εγγεγραμμένα, ε, υπάρχει θέμα επίλυσης των διαφορών, Υπάρχουν πλέον 300 εγγεγραμμένα συνδικάτα στη Βερμανία και ε, υπάρχουν και άλλα 500 τα οποία έχουν αιτήσει καθοδόν. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση να εισακούγεται η φωνή των εργατών ε, στη Βερμανία και αυτό φυσικά ενισχύεται και από το γεγονός ότι βλέπουμε αρκετές επιχειρήσεις πλέον ε, να εφαρμόζουν πολύ ε, μεγάλο ωράριο εργασίας, ε, ελάχιστους μισθούς και θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία πρέπει να βελτιωθούν ιδιαίτερα. Το ενδιαφέρον λοιπόν για τα συνδικάτα δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει και μας χαροποιεί το γεγονός ότι ήδη έχουν καταγραφεί τόσα πολλά συνδικάτα σε αρκετές επιχειρηματικούς κλάδους σε όλη τη Βυρμανία. Μας ανησυχεί λίγο το γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, διαπιστώνουμε ότι δημιουργούνται συνδικάτα στα οποία όμως διοικεί ουσιαστικά η διοίκηση μιας επιχείρησης ε, για να προσπαθήσουν να μειώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και να περιφεριοποιήσουν λίγο τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών ε, και συμφιλίωσης και διαιτησίας, ε, τα οποία είναι ευπρόσδεκτα φυσικά, αλλά είναι πολύ νέο το φαινόμενο και το κατά πόσον θα μπορέσει η κυβέρνηση να εφαρμόσει σωστά την νομοθεσία ε, είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να δούμε, αλλά υπάρχουν ε, κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν ε, και για θέματα ε, συμφιλίωσης και για θέματα διατησίας να κάνουν αυτό που πρέπει. Το, η Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, αυτό το οποίο θα ήθελε να δει ως απάντηση, ε, και νομίζω ότι η επαναφορά των δασμολογικών προτιμήσεων στο σύστημα γενετευμένων προτιμήσεων είναι μια καλή ευκαιρία, είναι να δούμε κατά πόσον μπορούμε να προχωρήσουμε τα θέματα αυτά με τη Βυρμανία. Η Επίτροπη Άστον και Ντεχούκτ φέτος μας είπαν ότι ε, θα πρέπει να γίνουν υπεύθυνε επενδύσεις, γιατί αυτές είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ε, ανασύστασης της χώρας. Και αυτό φυσικά αφορά και το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Και στις αρχές του έτους είχαμε ακούσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη Βυρμανία θα πρέπει να εφαρμόζουν τα υψηλά πρότυπα κεραιότητας ε, και αναφέρθηκαν και στις κατευθυντήρες γραμμές στο ΩΣΑ για τις επιχειρήσεις ε, και γενικότερα άλλα πρότυπα για τις επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η σωστή άγουσα φυσικά, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και όχι μόνο κάποιες ε, προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, πρόσφατα εξέδωσαν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ε, για την αποκάλυψη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βιρμανία. Θεωρούμε ότι αυτές δεν πηγαίνουν μέχρι εκεί που θα έπρεπε. Επιτρέπουν βέβαια την ε, αποκάλυψη πληρωμών προς την κυβέρνηση, ε, μια διαδικασία ε, screening για όσους ασχολούνται με θέματα φυσικού αερίου στη Βερμανία και ζητούνται από όσους έχουν πολιτικές δέουσας επιμέλειας να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες αυτές προς το ευρύτερο κοινό, να κοινοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Ε, Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι θα μπορούσε να πάει έτσι περαιτέρω. Θα θέλαμε να δούμε κάτι πολύ πιο εύρωστο, ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι παράλληλο με την ε, εφαρμογή εκ νέου των δεσμολογικών προτιμήσεων και να θεωρούνται όλα αυτά προϋπόθεση συνεργασίας με τη Βερμανία Να υπάρχει δέους επιμέλεια, να υπάρχει έλεγχος για τα θέματα αυτά και αν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις θα πρέπει μέσω δέουσας επιμέλειας να εξετάζονται όλα αυτά και να δημοσιοποιούνται ε, οι αλυσίδε προμηθειών στη Βυρμανία, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να υπάρχει και ευθύνη και λογοδοσία όσων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στη Βερμανία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η Βυρμανία εξακολουθεί να είναι ε, σε ε, επικίνδυνο επενδυτικό περιβάλλον, όχι μόνο το, λόγω των προβλημάτων που εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά και γιατί υπάρχουν ε, και μία σειρά από άλλες πολύ σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, θέματα κατάσχεσης γεών, για παράδειγμα, ε, θέματα τα οποία έχει καταγγείλει ο εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών στην πιο πρόσφατη έκθεσή του πριν από ένα μήνα, άλλωστε κατήγγειλε τα φαινόμενα αυτά στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ολοκληρώνοντα θα ήθελα να κάνω μία έκκληση να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει λίγο παραπέρα από αυτό που έχει κάνουν, κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και η Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικάτων προφανώ και θα βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί και θα διευκολύνει την όλη διαδικασία στη Γερμανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον εισηγητή μας, Dave Martin. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο προλαλήσαντες για την πολύ σαφής ε, παρουσίαση εισηγήσεις τους. Είναι σαφές ότι ο δρόμος ακόμα είναι πάρα πολύ μακρύς και τα πράγματα εξελίσσονται. Με ανησυχεί βέβαια ο τρόπος με τον οποίο όλοι έτρεξαν και αναγνώρισαν ε, το καθεστώς στη Βυρμανία, έτσι, με υπερβολική ταχύτητα. Όμως όσον αφορά το προτιμησιακό καθεστώς πιστεύω ότι είναι σωστό να ανασταλούν επί τη βάση του προβλήματος για την ε, καταναγκαστική εργασία. Υπήρχαν βάσιμες αντιρρήσεις για τη συνέχιση του συστήματος και είναι σωστό να δεχτούμε ότι το, τώρα θα πρέπει να ξαναξεκινήσει τη λειτουργία του το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων το 2013, δεδομένου ότι έχουμε ένα νέο σύστημα που θα τεθεί ενισχύ το 2014. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βάλουμε οποιοδήποτε όρους και να το συσχετίσουμε το καθεστώς αυτό των δασμολογικών προτιμήσεων, αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε την εξέλιξη, τις θετικές εξελίξεις, να ζητήσουμε την εφαρμογή νομικών μέτρων, να, ε, να πιέσουμε τους επενδυτές που επενδύουν αυτή τη στιγμή στη Βυρμανία να είναι σαφείς και ξεκάθαροι ως προς τους στόχους τους και να αποδείξουν ότι οι επενδύσεις τους ωφελούν τη χώρα και τον πληθυσμό. Μπορούμε λοιπόν να πιέσουμε για πολλά πράγματα, πολλά μέτρα, να ζητήσουμε την ελευθερία ε, συνε, συνελεύσεων, ε, να, την ελευθεροτυπία και πολλά άλλα πράγματα τα οποία ακόμα υπολείπονται. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο ο τύπος ε, αλλά το αποτέλεσμα και όσον ακόμα παραμένει η καταναγκαστική εργασία μια πραγματικότητα ε, το πρόβλημα θα συνεχιστεί και για το 2014 οπότε θα παραβιάζονται οι κατευθυντήρες γραμμές μας όταν ο πρόεδρος ε, Μπαρόσο πήγε στη Ραγκούν στην πρωτεύουσα για να συζητήσει για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, έθεσε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζήτησε ε, από τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών να παρακολουθήσουν και να ενημερώνουν για τις αλλαγές. Για να μην ακρηγορήσω, πιστεύω ότι η Βυρμανία έχει κάνει τα πρώτα βήματα προς θετική κατεύθυνση τα πρώτα διστακτικά, διστακτικά βήματα πρέπει να τους, να τους ενισχύσουμε, πρέπει να τους βοηθήσουμε μέσω του καθεστώτος ε, γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, αλλά να παραμείνει πάρα πολύ στενή η εποπτεία μας για τις εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Εγώ πιστεύω ότι και ε, οι νομικές διατάξεις και τα τυπικά ε, ε, αιτιολογικά ισχύουν, είναι σαφέστατα. Υπήρχαν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους αναστάλει το καθεστώς προσωρινά και βεβαίως πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση της Κομισιόν για την εκτέλεση των νομικών υποχρέωσεων, αλλά όχι μόνο σαν αφορά την νομική πτυχή, ε, πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε αφενός τις βελτιώσεις, την πρόοδο γενικά και όχι μόνο να εστιάσουμε στο πρόβλημα της καταναγκαστικής εργασίας και για πολιτικούς λόγους πρέπει, έχει μεγάλη σημασία να δείξουμε ότι εμένουμε στη θέση μας όταν θα εισαχθεί το νέο σύστημα GSP και ότι αποφασίσουμε για μία κατάσταση που υπάρχει, αν αλλάξει η πραγματικότητα, τότε θα μεταβάλουμε και εμείς την προσέγγιση μας. Αυτό δεν σημαίνει, όπως είπε και ο Ντέιβιτ, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στη Βυρμανία. βεβαίω υπάρχουν. Και προβλήματα υπάρχουν με πολλές από τις ε, χώρες της ε, ε, αναγκαστικές γης και πολλά άλλα προβλήματα. Ε, δεν πιστεύω όμως ότι η επιμέρους επίλυση ορισμένων προβλημάτων είναι ο μόνος λόγος για την ε, επαναφορά των δασμολογικών προτιμήσεων. Η Βιρμανία δεν είναι Νορβηγία, ούτε θα γίνει ποτέ Νορβηγία. Αλλά πιστεύω ότι είναι σωστή η κατεύθυνση της ε, ε αποκατάστασης Εάν το νέο σύστημα, όταν το νέο σύστημα ισχύσει, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται επί τη βάση του κανονισμού που αφορά αυτή τη χώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό που είναι λογικό από πλευράς Επιτροπής μας είναι να υιοθετήσουμε τη θέση της Κομισιόν. Ο Νίκολαϊ, ευχαριστώ Πρόεδρε, και εγώ συμφωνώ με τον Κρίστοφερ. Πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι σωστή. Αναφερθήκατε σε συντομία ε, ε, στις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών και τι προσπαθούν να επιτύχουν στη Βυρμανία. Πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί ένας συντονισμός με άλλα κράτη επενδυτών με την Ιαπωνία, παραδείγματο χάρη και άλλες χώρες που επενδύουν, για να μπορεί να γίνει μια κοινή προσέγγιση σε αυτή την πολιτική. Ο Ρόμπερ Στέρντι, ο οποίος είναι εδώ, ναι, συμφωνώ και εγώ με τον Κρίστοφερ. Είναι σωστό να υιοθετήσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Αλλά όσον αφορά τον, αυτά που είπε ο κύριος Ταπιόλα και ο κύριος Μπέργκ, ε, η έλλειψη άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βερμανία. Εάν υιοθετήσουμε αυτή την πρόταση της Κομισιόν θα δώσουμε ένα έναυσμα, θα ενθαρρύνουμε τις άμεσες ξε, ξένες επενδύσεις στη χώρα. Γιατί είναι σημαντικό ότι να υπάρχει σταθερότητα για επενδυτές. Όλοι οι επενδυτές θέλουν ένα σταθερό καθεστώς. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Αργεντινή, αλλιώ δεν θα επενδύσουν, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Αν θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε, ε, Υιοθετώντα αυτή την πρόταση θα βοηθήσει, θα τους ενθαρρύνει ο πρόεδρος. Α απαντηθεί αυτή η ερώτηση αργότερα, τη σημειώσαμε. Ας ακούσουμε τη Φρανσίσκα Κέλλερ τώρα. Ευχαριστώ. Και εμείς έχουμε δύο επιφυλάξεις γενικής φύσεως. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ήδη αναφέρθηκαν, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και θα έλεγα τα προβλήματα αυξάνονται όσον αφορά τις μειονότητες, τη μουσουλμανική μειονότητα στο Μιανμάρ, εκεί οξύνονται τα προβλήματα. Χρειάζεται βελτίωση και βεβαίως υπάρχουν και συγκεκριμένοι όροι που πρέπει να τηρηθούν. Μία άλλη ανησυχία που έχουμε είναι ότι ναι μεν να βοηθήσουμε το Μιανμάρ να αναπτυχθεί με δημοκρατικό τρόπο και να αναπτύξει και την οικονομία του. Και κατανοώ ότι υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις, ορισμένα προγράμματα που έχουν μελετηθεί μαζί με το, τις αρχές της χώρας. Διότι αν θέλετε να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του τοπικού εμπορίου, όχι μόνο στις εξαγωγές και στην, ε, ε, σε μια πολυδιάστατη οικονομία, όχι μόνο εξαγωγική. Τώρα, αν δούμε τι έχει γίνει τους τελευταίους μήνες στο Μιανμάρ, όλοι τρέχουν και δεν προλαβαίνουν. Πηγαίνουν στη χώρα γρήγορα να προλάβουν ένα μερίδιο της αγοράς, να εξασφαλίσουν συμβάσεις εξαγωγών πρώτων υλών, ενώ σύμφωνα με τις συνθήκες μας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει την ανάπτυξη της χώρας, όπως ανέφερα, και όχι να βοηθήσει αυτόν τον αγώνα δρόμου που γίνεται για πρόσβαση στις πρώτες ύλες και σε συμβάσεις που αυτή τη στιγμή είναι διαφαινόμενη τάση. Η Αυστραλία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, οι Εμείς Πολιτείες έχουν, κάνουν αγώνα δρόμου. Ποιος θα προλάβει να κλείσει τις συμφωνίες. Και το, το θέμα είναι, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω μετά από την προσχώρηση στο σύστημα δασμολογικών προτιμήσεων τι προγραμματίζεται για αργότερα, δεν ξέρω τι ε, εμπορική πολιτική έχουμε υπόψη μας και τι είναι δυνατόν να γίνει ρεαλιστικά. Κάθε φορά που συνομιλώ με την Κομισιόν, μου λένε ότι ναι, έχουμε κάποια επόμενα βήματα, ε, δεν ξέρω ακριβώς βέβαια τι θα γίνουν στις εμπορικές μας σχέσεις, αλλά αυτή τη στιγμή σας είπα, δεν πρέπει εμείς να δώσουμε την εντύπωση ότι συμμετέχουμε στον αγώνα δρόμου εξασφάλισης πρώτων υλών και θα πρέπει να βοηθήσουμε γενικώ την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με όλους τους τρόπους. Ποιος Μέρφυ για την ΚΟΕ. Ε, η πράγματι αξίζει να θέσουμε το ερώτημα γιατί βιάζονται όλοι να πλησιάσουν την πορμά. Είναι λίγο ύποπτο. Σίγουρα δεν οφείλεται μόνο στην βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Αντιθέτως ότι σχετίζεται με οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα ιδιαίτερο της καπιταλιστική υπηρελιστικής ε, ε, Αμερικής των σε σχέση με την Κίνα βέβαια. Ε, γι' αυτό το λόγο όλοι βιάζονται να ανοίξουν αγορές, ε, να αποκτήσουν πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Ε, όλο αυτό έχει σχέση με τον εμπορικό πόλο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Οπότε μην ξεχνάμε το, την πρόληψη αυτής της πρότασης. Ασφαλώς καλωσορίζουμε την πλήρη απαγόρευση της καταγκαστικής εργασίας. Ε, αναγνωρίζουμε ότι έχει μειωθεί, παρόλο που δεν έχει εξαλειφθεί. Όμως θα πρέπει να συζητήσουμε γενικότερα το θέμα των, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Μιανμάρ. Ε, ασφαλώς και η Βερμανία δεν είναι Νορβηγία, αλλά με αυτόν τον τρόπο τα βάζουμε όλα κάτω από το χαλί, διότι στην Μιανμάρ υπάρχουν άνθρωποι, εργάτες, εργαζόμενοι κλπ. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να γνωρούμε και όλα τα υπόλοιπα πέραν της καταγκαστικής Ασίας. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πέρασε ένα νόμο τον Σεπτέμβριο για να ε, σταματήσουν οι εθνοτικές διαμάχες μεταξύ μουσουλμάνων και βουδιστών ε, που προκάλεσαν το θάνατο χιλιάδων κυρίως μουσουλμάνων ενώ εξανάγκασε σχεδόν 100.000 άτομα ε, να ε, μετακινηθούν και πολλές χιλιάδες να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Ε, όλα αυτά, όλη αυτή η βία οφείλεται στην πολυετή καταπίεση μειονοτήτων. Το κράτος πρέπει να πάρει θέση Και δεδομένου ιδιαίτερα ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει και το ίδιο συμμετάσχει σε εκδηλώσεις βίας. Και ε, ένα άλλο πρόσφατο θέμα, τέλος Νοεμβρίου, ίσως διαβάσατε την, τον, την διάλυση ε, κατασκηνώσεων καταβλισμών διαμαρτυρώμενων κατοικών, κατοίκων σε μια ε, περιοχή της χώρας, ε, διαλύθηκαν δια της βίας, έχουν δικαίωμα όμως να διαμαρτύρονται, ποτέ δεν ε, έχουν καταφέρει να το εξασκήσουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν, τραυμάτισαν τουλάχιστον 40 άτομα, είναι σοβαρή η κατάσταση, θα πρέπει όλα αυτά να τα θέτουμε, συμφωνώ με τον εκπρόσωπο της ITUC, που ανέφερε το θέμα του ρόλου των ευρωπαϊκών πολυεθνικών εταιριών. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε την δική του συμπεριφορά στην Μιανμάρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας ε, για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Δύο λεπτά στον καθένα. Το ερώτημα που ετέθη ήταν αν ε, θα ενθαρρυνθούν με αυτόν τον τρόπο ε, οι άμεσες ξένες επενδύσεις με την αναστολή της, ε, με την αναστολή της, ε, ε, των περιορισμών. Σίγουρα η μία αναστολή θα επηρέαζε τις επενδύσεις από τις ευρωπαϊκές χώρες, όχι όμως από τις άλλες χώρες. Και έχουμε δει τι κάνουν οι άλλες χώρες. Ε, δεν νομίζω ότι βιάζεται η Ευρώπη. Υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον για την Μιανμάρ. Οπότε σκεφτείτε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ε, για να έρθουμε σε επαφή, σε διάλογο με τους επενδυτές και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ο ILO ε, έχει εντολή να παρακολουθεί ε, τις ε, επιπτώσεις της εργασιακής σχέσης και θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τις επιπτώσεις αυτού του ανοίγματο εννοώ. Κάτι άλλο. Ένα σύντομο σχόλιο παρακαλώ. Αν η καταναγκαστική εργασία μπορούσε να εξαλειφθεί εν μία νυχτή, δεν θα χρειαζόμαστε ένα αδιαίτες πρόγραμμα. Uh, Για τις δύο ερωτήσει ε, να πω τα Με την απελευθέρωση των επενδύσεων και την άρση των εμπορικών φραγμών στι ε, στις Ηνωμένες δεν είδαμε ε, μια μεγάλη κατακόρυφη αύξηση των επενδύσεων από τις ΗΠΑ τουλάχιστον, ε, εξαιτία του ότι ε, υπάρχουν περιορισμοί, πρακτικοί περιορισμοί, για παράδειγμα σχεδόν όλες οι συναλλαγές γίνονται με ρευστό, δεν υπάρχει πίστοση. Ε, οπότε υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι πραγματικά εμποδίζουν την αύξηση των επενδύσεων ε, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ανεξαρτήτως στήματος γενικευμένων προτιμήσεων θα πρέπει να αρθούν και αυτοί οι περιορισμοί για να αυξηθούν οι επενδύσεις. Η Coca-Cola, η Pepsi και η General Electric νομίζω είναι οι μόνες τρεις ε, μεγάλες πολυεθνικές που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να μπουν στην αγορά της Μιανμάρ. Από την άλλη μεριά η Κίνα, η Κορέα, η Ταϊβάν, η Ιαπωνία κλπ. Ε, πενδύουν εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα, Σε ό,τι αφορά τι ΗΠΑ, οι ΗΠΑ προσπαθούν ε, να ε, προωθήσουν μια πολιτική δέουσας επιμέλειας και αποκάλυψης ε, της ταυτότητας των επιχειρήσεων. Έχουν ένα κατάλογο με φυσικά και νομικά πρόσφατα, τον οποίο διατηρεί το Υπουργείο Οικονομικών και ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών. Ε, είναι ένας κατάλογος επιχειρήσεων και πολιτών με τους οποίους και τις οποίες δεν επιτρέπεται η συνεργασία από πλευράς αμερικανικών επιχειρήσεων εξαιτία του ότι είναι παράνομες οργανώσεις, ε, διεφθαρμένες κλπ. Και πρόσφατα ε, προέκυψε και μια καινούργια υποχρέωση από πλευράς των επιχειρήσεων ε, ε, αν θέλουν να κάνουν κοινέ επιχειρήσει να συνεργαστούν ε, στον τομέα του πετρελαίου, ε, πρέπει να αποκαλύπτουν εγκαίρως αρκετά νωρίτερα ποιοι είναι οι συνεργάτες τους και διάφορα στοιχεία για αυτή τη συνεργασία. Αν μια εταιρεία έχει μια πολιτική, ακολουθεί μια πολιτική ε, δέουσα επιμέλεια, αυτή θα πρέπει να είναι δημόσια. Το ερώτημα βέβαια είναι το κατά πόσον υπάρχει μόνο πολιτική ή πράγματι επιδεικνύεται ιδέως επιμέλεια, διότι ε, γενικά ε, μέχρι τώρα δεν υπάρχει υποχρέωση αποκάλυψης, ε, δημοσίευσης του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Ε, και αυτό αποτελεί ένα κενό. Πρόεδρος, Κομισιόν, Φρανσίσκο Πέρεθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια διότι προφέρετε εξαιρετικά το αδύνατο να προφέρει κανείς όνομά μου. Ε, εμείς θα λάβουμε υπόψη φυσικά όλες σας τις συζητήσεις. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα fact sheet εδώ το οποίο διανύμαμε την περασμένη εβδομάδα που απαντά και μια σειρά από ερωτήσεις ε, που θέσατε σήμερα. Να επισημάνω ένα-δυο σημεία βέβαια. Από ό,τι ακούσαμε το κοινό θέμα ε, είναι η νομική πτυχή του καταναγκαστικής εργασίας και την ανάγκη να έχουμε το σύστημα ε, προ... γενικευμένων προτιμήσεων χωρίς κανένα όρο, οποιαδήποτε μορφής όρους. Και φυσικά αυτό ε, να σας υπενθυμίσω ότι όταν, αν κάνουμε οτιδήποτε προς αυτή την κατάσταση, όχι μόνο θα δημιουργήσουμε κίνδυνο, αλλά θα δημιουργήσουμε και πρόβλημα με βάση τις αρχές του ΠΟΕ. Για να σας απαντήσω σε κάποιες από τις ανησυχίε, ε, είναι σημαντικό να σας πω ότι σε περίπτωση που αναστραφεί η πρόοδος και δεν αναφέρομαι μόνο στην καταναγκαστική εργασία, αλλά στις συμβάσεις εργασίας και τις συμβάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, έχουμε δικαίωμα βάσει του νο... της νομοθεσίας μας να αποσύρουμε και πάλι το σύστημα ε, γενικευμένων προτιμήσεων. Αλλά ε, η λύση λοιπόν υπάρχει. Αλλά όπως είπε και ο εισηγητής, από 1η Ιανουαρίου του 2014 θα μπορούμε να το κάνουμε και επί τη βάση αποδείξεων που θα δίνονται από αξιόπιστες πηγές, ε, ακόμα και εσά του ίδιους κυρίες και κύριοι. Επομένως ο μηχανισμός υπάρχει. Ε, Κατά τα άλλα, αναφέρθηκαν κάποιοι στόχοι. Φυσικά θεμητοί όλοι αυτοί οι στόχοι και συμφωνούμε επ' αυτού. Ε, το να υπάρχουν ε, αρχέ, υπεύθυνε επιχειρήσει και ούτω καθεξής. Αλλά σα παρακαλώ, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Η αίσθησή μας είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, αυτά όλα τα θέματα σε άλλες περιπτώσεις που είναι καλύτερο να γίνουν η συζήτηση και δεν θα πρέπει να ε, ξεχνούμε και τι σημαντική συνεισφορά μπορεί να κάνει το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων γιατί μπορούμε να έχουμε πρόοδο μέσω αυξημένων πόρων. Να σας ε, πω επίσης και νομίζω ότι αυτό είναι και μια πολύ σημαντική ερώτηση αν η Επιτροπή έχει ένα ε, βασικό σχέδιο, ένα master plan. Δεν έχουμε πάντα master plan γιατί μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Υπάρχει όμως μια ολιστική προσέγγιση και η ολιστική μας προσέγγιση είναι σίγουρα μια προσέγγιση που βασίζεται και στην ε, ανάπτυξη υποστήριξη. Στο fact sheet προσπαθούμε να σας δώσουμε κάποια καλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, καλή διακυβέρνηση και ανθρώπινα ε, δικαιώματα θα είναι οριζόντια συνιστό σα ε, στο σύστημα τεχνικής συνδρομής το οποίο προετοιμάζουμε, επομένως τα λαμβάνουμε υπόψη. Επίσης, να υπογραμμίσω ότι Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία απασχολούν ε, το σύστημα, ε, την συνεργασία ε, και όχι το σύστημα γενικευμένων προτιμώσεων. Από το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είπε ότι θα παρακολουθεί τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις για να τηρούν κάποιες αρχές και κοιτάμε να δούμε κατά πόσον εφαρμόζονται οι αρχές αυτές του CSR και στον τομέα του φυσικού αερίου, στο ΛΑΝΚ και όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια ενός τριμερούς διαλόγου που αφορά τις εκθέσεις, τη βελτίωση των εκθέσεων των επιχειρήσεων για περιβαλλοντικές και κοινωνικές πληροφορίες, καθώς επίσης και μία ε, πρόταση για δημοσιοποίηση πληρωμών προς κυβερνήσεις, ε, τα οποία όλα αυτά αφορούν τη Μιανμάρ. Δεν έχουμε λοιπόν ένα master plan, αλλά μια ολιστική προσέγγιση για να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα θέματα, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο Όπως είπε και η Αν Σουκέν και θα παραθέσω αυτό που είπε, η άρση ή αναστολή των ε, κυρώσεων και η ε, επαναφορά του συστήματος γενικευμένων προετοιμήσεων δίνει μια δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης που θα πρέπει να αποτελεί ικανή και αναγκαία ε, συνθήκη της δημοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ευημερίας της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν με το θέμα αυτό, ο Ντέιβιτ Μάρτιν, ο εισηγητή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συνεχίσω από κάτι που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είμαστε σαφείς για τη συνεισφορά μου. Είπα ότι έχουμε μια δυνατότητα Από νομική σκοπιά λίγα μπορούμε να κάνουμε παρά μόνο να επαναφέρουμε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ε, και αυτό φυσικά λαμβάνοντα υπόψη και τι αλλαγέ ε, που γίνονται. Συμφωνώ μεν για αυτό που είπατε για του όρου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, πρέπει να σχολιάσουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για τις δράσεις τις οποίες σκοπεύετε να αναλάβετε πέραν του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Δεν ε, υπάρχει λόγος να μην αναφέρουμε στο ψήφισμά μας και άλλα πράγματα τα οποία αφορούν την κατάσταση στη Βερμανία. Ιδίω στο θέμα της εταιρική κοινωνικής ευθύνη και δεν υπάρχει και λόγο λόγος να μην επιμείνουμε ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Μπαρόζο τα ευρωπαϊκά κονδύλια λοιπόν που δίνουμε προς τη Βυρμανία και καλά κάνουμε και τα δίνουμε, είναι όμως χρήματα τα οποία δίνονται στη Βυρμανία και γιατί να μην χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρύνουμε τη βελτίωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας, να μην ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της πολιτικής διαδικασίας, να παρακολουθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την οδηγία για τη διαφάνεια, για να ε, λαμβάνονται οι πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται στη Βυρμανία όπως και σε άλλες χώρες, και να λάβουμε υπόψη και θέματα μειονοτήτων και να αναβαθμίσουμε τη σχέση μας με τη Βερμανία. Για να, να βαθμιστεί αυτή η σχέση θα πρέπει να υπάρχουν και ψηλέ προδιαγραφές από πλευρά της χώρας. Ναι, μεν δεν μπορούμε να τα θέσουμε ως όρους για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, αλλά θεωρώ ότι είναι προαπαιτούμενο το Κοινοβούλιο να θέσει όλους αυτούς τους όρους ε, και να τους αναφέρει για την ε, ε, επαναφορά του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων να σας πω ότι θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε το θέμα μέχρι το τέλος του 2013 και ε, να δούμε και τι γίνεται και με τη νέα γενεά του συστήματος γενικευμένων προεδρυμίσεων μετά το 2014. Συμφωνώ βέβαια με τα όσα είπε ο μιλητής από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ότι ωραίο θα ήταν να γίνουν τα πράγματα έτσι, αλλά όλα χρειάζονται χρόνο. Αυτό που θέλουμε είναι να διαπιστώσουμε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος και να διασφαλίσουμε ότι οι και αλλαγέ στην νομοθεσία αντανακλούν την πραγματικότητα στη χώρα. Διότι ξέρουμε ότι σε κάποιε περιπτώσει δεν συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχουν χώρες με τέλεια συντάγματα και ε, πρότυπα νόμου ε, και η κατάσταση στην πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Στη Μιανμάρ λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθούμε για να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνουν οι αλλαγέ. Και πέραν αυτού κύριε Πρόεδρε, εγώ προτείνω για να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι ο συζητητής θα κάνω προτάσεις για να αλλάξει νομοθεσία, αλλά θα ήθελα με την άδειά σας να ετοιμάσω και ένα σχέδιο που θα συνοδεύει το ψήφισμα με κάποιες προτάσεις για να τις λάβετε υπόψη για τα υπόλοιπα θέματα. Ευχαριστώ. Ωραία, εντάξει, σημειώσαμε τις προθέσεις σας και την προσέγγιση σας. Χρονοδιάγραμμα. Ε, συζήτηση σχεδίου γνωμοδότησης τον ερχόμενο Φεβρουάριο, του σχεδίου έκθεσης, ε, τον ερχόμενο Φεβρουάριο στην τακτική συνεδρίαση και αυτό ήταν το τελευταίο θέμα πριν από τη συνεδρίαση των συντονιστών. Ε, είμαστε 15 λεπτά νωρίτερα από το πρόγραμμά μας και θέλω να σας ρωτήσω εάν θέλετε να αρχίσουμε τώρα. Προτείνω να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα για να δώσουμε την ευκαιρία να έρθουν οι συγητές που λείπουν. Αλλά εγώ βλέπω ότι σχεδόν όλοι είναι παρόντες εκτός των πρασίνων. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε ένα διάλειμμα πέντε λεπτών και να συνεχίσουμε. Με... Αφού όσοι δεν έχουν θέση στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών αποχωρήσουν από την αίθουσα. Βοηθή κλπ.